Przewodniczący! Hello. Good morning, colleagues. Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζει η συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα της ε, συνεδρίασής μας είναι η έκθεση του κυρίου Σαλβατόρ Γκαρίκα Πολέτο σχετικά με την επένδυση στο μέλλον. Είναι ένα νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. Το λόγο θα πάρει καταρχήν ο ίδιος ο εισηγητής. Κύριε Σαλβαδόρ Γκαρίγα Πολέτο, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επιτρόπε Λεβαντόφσκι, συνάδελφοι, εδώ και 23 χρόνια εκδίδουμε δημοσιονομικέ προοπτικέ σε τέσσερι διαφορετικέ περιόδου που έχουν ε, συνεισφέρει στην ε, εξέλιξη των δαπανών και των εσόδων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια ύπαρξη των δημοσιονομικών προοπτικών ε, κατέστησε δυνατή την εξέλιξη και εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Συνεπώ, η συζήτηση αυτή και η μεταγενέστερη ψηφοφορία έχει σημασία για τα οικονομικά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίρνει πρωτοβουλία ε, στον πολιτική πρωτοβουλία στον, ε, υποβάλλοντας μια πρόταση και η Κομισιό και το Συμβούλιο θα αντιδράσουν σε αυτή την πρόταση. Έχουμε έτοιμη μια πρόταση ε, συνενετική και συνεργατική. 1.100 τροπολογίες, ένας χρόνος εργασίας, 120 συμβαστικές προτάσεις, 11 ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές και 10 εθνικά κοινοβούλια συνεισέφεραν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους εργάστηκαν αυτό το χρόνο για να γίνει δυνατή αυτή η έκθεση. Ε, διοργανική συμφωνία. Ο κύριος ε, Ντρόμπα Μπαρόσο ε, και ο Επίτροπος κύριος Λεβαντόφσκι συνεργάστηκαν πάρα πολύ μαζί μας. Ελπίζουμε ότι η δική τους πρόταση που θα εκδοθεί στις 29 Ιουνίου θα είναι συμβατή με τις δικές μας προτάσεις. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με, την, με περισσότερη Ευρώπη και μικρότερο προϋπολογισμό. Όχι πια. Θέλουμε να τελειώσουμε, να ε, να σταματήσει πια η ανάληψη ε, δεσμεύσεων χωρίς οικονομική υποστήριξη. Ε, έχουμε αναλάβει ήδη δεσμεύσεις ε, για την Ευρώπη του 2020 και δεν θέλουμε αυτή να, γίνει, να, έχει, να έχει τη μοίρα που είχε η στρατηγική της Λισαβόνας. Γι' αυτό το λόγο η στρατηγική 2020 είναι ο βασικός άξονας των δημοσιονομικών προοπτικών. Πιστεύουμε στην αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών δαπανών. Ένα ευρώ του ευρωπαϊκού προπολογισμού είναι πιο αποτελεσματικό και ε, από ε, το 1 ευρώ στους 27 εθνικούς προϋπολογισμούς. Γι' αυτό το λόγο ε, η αρχή μας είναι η προσθέμενη αξία, ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και πιστεύουμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ζητούμε αυτό να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι δυνατόν να κατανοήσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική χωρί επαρκή χρηματοδότηση στην αγροτική πολιτική και την πολιτική συνοχή. Γι' αυτό το λόγο ζητούμε από το Συμβούλιο να διατηρήσει το επίπεδο των δαπανών και στις δύο αυτές πολιτικές και μετά το 2013. Έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία, επενδύσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας, κλιματική αλλαγή και παιδεία είναι μερικές από τις προτεραιότητες που θα πρέπει να καλύψει ο προπολογισμό. Πιστεύουμε ότι η μείωση του κοινοτικού προπολογισμού δεν είναι βιώσιμη διέξοδος για μας που πιστεύουμε στην ανταγωνιστική Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ένα, μια αύξηση τουλάχιστον 5% στα, στις ε, δαπάνες για τις δημοσιονομικές προοπτικές και αυτό είναι το ελάχιστο που είναι απαραίτητο για να καλύψουμε τις ε, νέες προτεραιότητες και τις παραδοσιακές μας πολιτικές. Αυτό το 5% αποτελεί δείγμα πολιτικού ρεαλισμού και θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την κατοπινή ε, διαπραγμάτευση μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ε, και βέβαια χρειαζόμαστε και ένα καινούριο σύστημα ιδίων πόρων όπως συμφωνήσαμε. Ίσως είναι ε, ε, ε δύσκολη στιγμή εξαιτία ε, των μνημονίων και της κρίσης. Αλλά όλοι όσοι πιστεύουμε ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό είναι το πιο κατάλληλο εργαλείο έτσι ώστε τα 27 κράτη-μέλη να γίνουν πραγματική ένωση ε, θα αναλάβουμε τις ευθύνε μας ενώπιον αυτού, αυτού, αυτής της πρόκλησης. στη συζήτηση θα δούμε ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά σημεία του υπερπολισμού. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ε, την συνένεση, την ομοφωνία στο Κοινοβούλιο, αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ τι πολιτικέ ομάδε για τη γενναιοδορία με την οποία αντιμετώπισαν όλη αυτή τη διαδικασία. Χάρη σε αυτέ τι ομάδε. η τελική έκθεση είναι πολύ καλύτερη από ότι ε, η αρχική μου πρόταση και από ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσα να έχω πετύχει μόνο μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ συνάδελφε ο πρόεδρος κύριος Τζόζεφ Ντόλ. Κύριε πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, να πάρω μια ανάσα. Η κρίση του ευρώ, του δημόσιου χρέους, απαιτεί ευρωπαϊκές και όχι εθνικές λύσεις. Αυτό είναι το μήνυμα που μαζί με την Επιτροπή του Χωσέ Μανουέλ Μαρότζο έχει στείλει στο Κοινοβούλιο μας εδώ και μήνες. Δηλαδή, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση συνεπά... Ε, ευρωπαϊκή λύση, συνεπάγεται ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες λύσεις της πραγματικότητας της Ευρώπης και στην οτροπία. Και θέτω το ερώτημα προς το Συμβούλιο. Η Ευρώπη της δεκαετίας του 20 είναι του 2020 θα είναι η ίδια με την Ευρώπη του προηγούμενου αιώνα. Η ανάπτυξη, η θέση της Ευρώπης στον κόσμο συγκρίνονται. Φυσικά όχι. Σήμερα η Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη των ιδρυτών της. Άλλαξε και θα ήταν ανεύθυνο να μην φανούν αυτές οι αλλαγές στον τρόπο που χρηματοδοτείται η Ένωση, δηλαδή που έχει συλληφθεί. Κύριε Πρόεδρε, θα δώσω το λόγο στον Μάρτιν Σούλτ. Ζητώ συγγνώμη, θα πάρω το λόγο μετά, αν δεν έχετε αντίρρηση. Έτρεξα πάρα πολύ γρήγορα και πιέστηκα. Εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Σούλτ. Έχετε το λόγο, κύριε Σούλτ. Αλλά θα πάρω όμως και το χρόνο γόρευσης που απομένει, κανένα πρόβλημα. Ε, που σημαίνει ότι γιατί όχι να εκπροσωπήσω και το ΕΛΚ, να μιλήσω και εκ μέρους του ΕΛΚ. Πολύ ωραία. Ε, καταρχήν, ε, Πρόεδρε, θέλω να πω ότι ένα θερμό ευχαριστώ στον εισηγητή και στους συναδέλφους της ε, προσωρινής της ad hoc επιτροπής ε, οι οποίοι κατά την άποψή μου παρουσίασαν ένα θαυμάσιο έργο. Σπάνια πρέπει να πω έχω δει μια τόσο ισόρροπη και λογική έκθεση ε, όπως είναι αυτή που την κατέθεσε η ad hoc επιτροπή, η ΣΟΥΡΕ. Όσον αφορά τώρα το θέμα των μελλοντικών δημοσιονομικών προοπτικών και τη διαμόρφωσή του κύριε και κύριοι, εκεί ακριβώ φαίνεται τι είδου Ευρώπη επιθυμούμε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένας προϋπολογισμός για τα επόμενα έτη, ένας προϋπολογισμός ο οποίος θα αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες των κρατών μελών, αλλά όχι μόνο αυτών, αλλά και των προέδρων, αρχηγών, κρατών και κυβερνήσεων και των πολιτών μας. Πίσω λοιπόν από αυτές τις ε, δίθεν συζητήσεις ε, για, τα, ε, για τους δεκαδικούς αριθμούς, επί της ουσίας πρόκειται για την κατεύθυνση που θα λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τα επόμενα δέκα χρόνια. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα κατατίθενται νέες προτάσεις. Τι υποτίθεται ότι πρέπει να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι πρέπει να προσφέρει, γιατί είδου καθήκοντα πρέπει να προετοιμαστεί και παράλληλα διαπιστώνουμε ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο είναι απαραίτητο για να γίνουν όλα αυτά, κατ' ουσίαν δεν υφίσταται. Αν όμως επιθυμούμε να εκχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερες αρμοδιότητες και αν περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει φιλόδοξα προγράμματα από την άλλη πλευρά όμως προβαίνει σε περικοπές τούτο σημαίνει ότι έχουμε ξεκινήσει το δρόμο της μη αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματο χάρη στην πολιτική συνοχή. Αυτό ισχύει. Ισχύει ότι δεν υπάρχει πλέον αλληλεγγύη, μια αλληλεγγύη η οποία πραγματικά ε, πλέον διακυβεύεται. Αυτή η αλληλεγγύη πλέον πίσταται ε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει βέβαια και η Ευρώπη την οποία οραματίζεται ο κύριος Κάμερον, η Ευρώπη την οποία επιθυμεί η Ολλανδική κυβέρνηση ή τουλάχιστον οι ευρωβουλευτές που στηρίζουν την κυβέρνηση αυτή. Δηλαδή η Ευρώπη των όλο και περισσότερων περικοπών, μια Ευρώπη της όλο και μεγαλύτερης απόσυρσης από τη διαδικασία ανάπτυξης, ανάπτυξη, μια Ευρώπη τη επανεθνικοποίηση. Βεβαίω και υπάρχουν κάποιοι που επιθυμούν μια τέτοια Ευρώπη. Πρέπει όμω να πούμε ότι η Ευρώπη είναι και η απάντηση που θα δώσουμε εμεί κατά τον 21ο αιώνα στι οικολογικέ, οικονομικέ, δημοσιονομικέ, νομισματικέ και μεταναστευτικές προκλήσεις και όλα αυτά ε, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Έχουμε λοιπόν δύο εναλλακτικές λύσεις. Βεβαίως ε, μπορούμε αν θέλετε να κατακαιρματιστούμε σε μικρές οντότητες. Θα έχουμε τη Γερμανία με 82 εκατομμύρια και θα φτάσουμε και μέχρι τη Μάλτα με 360.000 κατοίκους. Και ο καθένας ε, μόνος του θα προσπαθεί, ε, τότε και η Ευρώπη θα χάσει τη σημασία της γιατί μια χώρα με 82 εκατομμύρια όπως αυτή που εκπροσωπώ εγώ, μα μια τέτοια χώρα στο πλαίσιο της, του διπυρωτικού ανταγωνισμού δεν θα μπορεί και αυτή να ανταπεξέλθει. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι τα 500 εκατομμύρια. Τα 500 εκατομμύρια σε μια κοινότητα. Χρειαζόμαστε τα 27 κράτη και αν τα διαθέτουμε αυτά τότε είμαστε ισχυροί. Αυτό ακριβώς λοιπόν σημαίνει ότι κατά τα επόμενα 7 έτη στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προοπτικής μέχρι το 2020 πρέπει να έχουμε κατά νου αυτά που σας είπα. Το σχέδιο που έχει κατατεθεί είναι ικανοποιητικό και επιθυμώ όλα αυτά να φανούν και κατά διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Μια συνεργασία που θα επηρεάσει την Ευρώπη, ε, τα κράτη ε, θα διαπραγματεύονται, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης για να ορίσουν το δημοσιονομικό μέλλον της Ευρώπης. Δεν μπορούμε να λέμε ότι επιθυμούμε να υπάρχει ένα πρόγραμμα Marshall για την Μεσόγειο, να βοηθήσουμε τις δημοκρατίες της Βόρειας Αφρικής, παράλληλα όμως να προβαίνουμε σε περικοπές του ευρωπαϊκού προπλογισμού. Δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση με 0,8 του ΑΕΠ και ε, ως πρώτη κυβέρνηση η Γερμανία να ζητάει αποζημιώσεις ε, όταν πλήττονται οι αγρότες της ε, από το E. το βακτήριο E. Το ίδιο έκανε και η Ολλανδία. Βεβαίως και πρέπει να βοηθήσουμε τους γεωργούς. Όμως για να τα πράξουμε όλα αυτά χρειαζόμαστε έναν ισόρροπο, λογικό, προϋπολογισμό, μακρόπνο προϋπολογισμό, ακριβώς όπως αναφέρεται στην έκθεση που έχει κατατεθεί. Λοιπόν, είστε, έτοι, είστε έτοιμος κύριε Πρόεδρε να απαντήσετε στην ερώτηση της ε, μπλε, μιας μπλε κάρτας. Λοιπόν, κύριε Χάρτονγκ. Uh, working? Okay. Dank u wel, voorzitter. Ik zou mijn gewaardeerde collega eh, willen vragen. Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τον συνάδελφο γιατί αντέδρασε αρνητικά στη θέση που έλαβε η Ολλανδική κυβέρνηση. Και σας ερωτώ συνάδελφε, το δημοκρατικό δικαίωμα των κρατών μελών να έχουν δική της άποψη και να την παρουσιάζουν αυτοί στους πολίτες τους, εσείς το αναγνωρίζετε ή όχι. Αγαπητέ συνάδελφα, μα προφανώς και το αναγνωρίζω αυτό το δικαίωμα. Μόνο που υποθέτω και θέλω να ελπίζω και εσείς να αναγνωρίζετε το δικαίωμα των υπολείπων να μην ε, υποκλίνονται όλοι ε, στην θέση της ε, Ολλανδικής κυβέρνησης αλλά να μπορεί να γίνεται μια συζήτηση στο πλαίσιο μιας ελεύθερης δημοκρατίας. Βεβαίως έχω και σεβασμό για τον κύριο Ρούντε ο οποίος είναι υπέρ της αύξησης του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 2,7% και χαίρομαι που με ακούσατε πολύ προσεκτικά γιατί σε αυτό το κοινοβούλιο οι θέσεις όλων των κυβερνήσεων κυβερνήσεων τα ανοιχτά. Κατόπιν τούτο δεν κατάλαβα ακριβώ τι θέλατε ε, από μένα, γιατί κάνατε αυτή την ερώτηση. Αλλά νομίζω υπενήσεστε ότι κι εσεί ε, στρατεύεστε και δεσμεύεστε στα δημοκρατικά δικαιώματα και, εν πάση περιπτώσει, καλό αυτό. Πρόοδο απαιτεί, αποτελεί. Ο κύριος Γκί Φερχόφστατ, πρόεδρος των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, έχω εδώ την επιστολή του εκπροσώπου της ε, κυβερνήσεως της αυτής μεγαλειότητας για την έκθεση Σούρα και λέει η επιστολή η κυβέρνηση αυτής μεγαλειότητας είναι απογοητευμένη από το σχέδιο έκθεσης ΣΟΥΡ. Δηλαδή, το σχέδιο έκθεσης ΣΟΥΡ είναι εξαιρετικό. Αυτό σημαίνει αυτή η επιστολή. Πρέπει να σας πω πέρα από τα τρία-τέσσερα λόγια αυτά, ότι η κυβέρνηση, δηλαδή ότι η κυβέρνηση της αυτής μεγαλειότητας είναι απογοητευμένη από την έκθεση. ότι η υπόλοιπη επιστολή αποτελεί πρόκληση προ την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι... Αυτό που συγκεκριμένα λένε είναι ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει αύξηση του ε, πι και ότι πρέπει να μείνουμε στο παλιό. Το παλιό με τα ίδια νούμερα, τους ίδιους πόρους, τις ίδιες φυσικά μειώσεις και φυσικά τη μείωση για το Ηνωμένο Βασίλειο και δεν θα αλλάξει τίποτα. Φυσικά η κυβέρνηση αυτής της μεγαλειότητας είναι μια κυβέρνηση που θέλει να λαμβάνει αποφάσεις και να μεταρρυθμίσει το Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί λοιπόν πρέπει να μείνουμε στο παλιό πι. Θα συνεχίσουμε δηλαδή με τις παλιές πολιτικές. Θεωρώ κύριε Πρόεδρε ότι έχει φτάσει πλέον η στιγμή να πούμε στην κοινή γνώμη ότι με το να περιορίζουμε τον προπολογισμό του 1% της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα λύσουμε την δημοσιονομική εξυγίανση των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 1% αυτό είναι το 1,4 μόνο των συνολικών δαπανών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει κι άλλος τρόπος να κάνουμε οικονομίες και υπάρχουν άλλοι τρόποι να κάνουμε την κυβέρνηση αυτής τη αν θέλουν να κάνουν οικονομίες στον Βρετανικό δημόσιο τομέα θα το κάνουν αυξάνοντας το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι μπορούν να εξοικονομήσουν πόρους. Τρία παραδείγματα θα σα δώσω. Πρώτον, η εξωτερική πολιτική. Γνωρίζετε ότι κάποιοι έχουμε 28.000 ε, ε, ε, διπλωμάτες στην Ευρωπα... στην... Ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και 93.000 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ, γιατί δεν δουλεύουμε όλοι μαζί. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργαζόταν περισσότερο, άλλο το Ηνωμένο Βασίλειο μπορούσε να συνεργαστεί περισσότερο, θα έκαναν οικονομίε, θα είχαν λιγότερου διπλωμάτε. Υπάρχει το θέμα τη νομισματική πολιτική. 44.000 άτομα στην Ευρώπη είναι υπεύθυνα για την νομισματική τη πολιτική. 44.000 στι Ηνωμένε Πολιτείε 18.000 στο Federal Reserve Board. Δηλαδή το ένα τρίτο, τρεις φορές λιγότερους από αυτούς που έχουμε εμείς. Αν λοιπόν η Βρετανική κυβέρνηση θέλει να κάνει οικονομίες, ας μπει στο ευρώ, ας δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα εξοικονομήσει όλους αυτούς οι υπαλλήλου που δουλεύουν για τα νομισματικά στη Βρετανία. Και αν θέλει να κάνει οικονομίες στη Μεγάλη Βρετανία, ας το κάνει στον τομέα της έρευνας λέγοντας υπάρχουν τα ευρωπαϊκά, ε, η τα θα τα χρησιμοποιήσουμε και θα κάνουμε τεράστιες οικονομίες στον προπολογισμό μας». Αυτά είναι ως απάντηση στην κυβέρνηση αυτής της μεγαλειότητας, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ο κύριος Τζόσεφ Ντόλ, πρόεδρος του ΕΛΚ. Συγγνώμη, ήθελα να τρέξω. Νόμιζα ότι ήμουν 30 χρονών, αλλά θυμήθηκα ότι είμαι 60. Euh, Είχα ήδη ξεκινήσει λέγοντας ότι η, μια... η χρηματοδότηση στην Ευρώπη πρέπει να προσαρμοστεί στις καινούριες πραγματικότητες της Ευρώπης και στους στόχους. Και ήθελα επίσης να πω ότι η δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών δείχνει ε, ότι οι προοπτικές ε, ανάπτυξης Ευρώπης ε, είναι, κάτι, ε, είναι πολύ περισσότερες από αυτές που είχαν φανταστεί οι ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να αντικατοπτριστούν στον τρόπο που χρηματοδοτούμε την, την Ευρώπη. Είναι η, η Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου διεξήγαγε μαζί με την Επιτροπή των Προπολογισμών μια πολιτική συζήτηση εδώ και ένα χρόνο. Ε, συγχαίρω την Επιτροπή Σούρε και ζητώ αυτό το ευρωπαϊκό πνεύμα, το ε, οποίο χαρακτήρισε τις εργασίες της, ε, να χαρακτηρίσει και τις εργασίες, ε, τις υπόλοιπες εργασίες, εδώ στην Ολομέλεια, στο μέλλον. Η, το, η ομάδα μας ζητά από τα κράτη-μέλη να συμμετάσχουν χωρίς περιορισμούς, χωρίς προκαταβολικά να πούμε ότι μέχρι το 2020 θα πρέπει η Ευρωπαϊκή, ο προπολογισμό να μην σταθερό, να παγώσει. Χρειαζόμαστε περισσότερο ευρωπαϊκό προπολογισμό, μεγαλύτερο, για να ανακουφίσουμε τους εθνικούς προπολογισμού. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε ιδίου πόρους. Ο Ευρωπαϊκό προπολογισμό άλλωστε ήταν ε, πάντοτε ισοσκελισμένο αντίθετα με πολλού εθνικού προπολογισμού. Επίση σα υπενθυμίζω ότι πάνω από το 90% των δαπανών του ευρωπαϊκού προπολογισμού ευνοούν τα κράτη-μέλη γιατί είναι επενδύονται σε σχέδια που ευνοούν τα κράτη-μέλη. Και, ε, όταν περισσεύουν ε, ποσά επιστρέφονται στον, ε, στα κράτη-μέλη. Πώς μπορούν να μας χαρακτηρίσουν για κακούς διαχειριστές. Ας πούμε την αλήθεια. Ένα ευρώ που δαπανάτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ένα ευρώ που δαπανάτε σε ένα εθνικό ε, προπολογισμό. Γιατί εκεί χάνει ήδη 20 ως 30% της αξίας του για να επιστραφούν ή ε, ε, τα δάνεια τα οποία, στα οποία έχουν καταφύγει οι εθνικοί προπολογισμοί. Μετά, ε, έχουμε ε, μια... αν, δεν κάνουμε, αν δεν προσαρμοστούμε θα εξακολουθούν οι μεγάλοι μας εγκέφαλοι να φεύγουν στις ΗΠΑ και στην Κίνα. Οι χώρες μας θα είναι λιγότερο ανταγωνιστικές και θα χάσουμε το στίχημα της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η αλήθεια είναι ότι χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της Επιτροπής Συνοχής οι διαφορέ ανάμεσα σε πλούσιες και φτωχέ χώρε θα αυξηθούν. Η αλήθεια είναι ότι χωρί ευρωπαϊκή χρηματοδότηση η πολιτική τροφιμικής ασφάλεια, η ενεργειακή πολιτική και η πολιτική καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών δεν θα είναι στο ύψο των περιστάσεων και των φιλοδοξιών μα. Τέλο, η αλήθεια είναι ότι χωρί χωρίς ευρωπαϊκή ε, χρηματοδότηση τη εξωτερική πολιτική και τη πολιτική ασφάλεια, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει να μην βρίσκεται στο κέντρο τη παγκόσμια κακέρα. Βέβαια, δεν είναι όλα ζήτημα χρημάτων. Και ο τρόπος με τον οποίο θα αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτεί συγκεκριμένες προτεραιότητες θα είναι ε, ζωτική σημασία για την δυνατότητα της Ευρώπης να επηρεάζει τον κόσμο στο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, οι πολιτικές ομάδες ε, συμφωνούν μαζί μου. Γι' αυτό το λόγο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει από το Συμβούλιο να ε, ανεξετάσει τη θέση του σε ό,τι αφορά τι δημοσιονομικέ προσωπικέ. Αν είναι σοβαρό στην δηλωμένη επιθυμία του να δράσει υπέρ της ανάπτυξης θα πρέπει να ε, δώσει στον προϋπολογισμό τα κατάλληλα μέσα. Αν είναι εξίσου σοβαρό με την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, θα πρέπει να καταλάβει το Συμβούλιο ότι ε, το να δαπανούμε πιο αποτελεσματικά είναι καλύτερο από το να δαπανούμε λίγο. Και το να δαπανούμε από κοινού είναι πιο λογικό από το να κατακαιρματίζουμε τις δαπάνες μας σε εθνικό επίπεδο. Το σχέδιο αυτό είναι ε, φιλόδοξο για την Ευρώπη και έχει την υποστήριξη της ομάδας μας. Αυτή η ελπίδα, αυτή η φιλοδοξία είναι που θέλουμε να δειχθεί στους πολίτες μας. Γιατί οι πολίτες μας στους δρόμους της Μαδρίτης και της ε, Αθήνας, ε, στο, τη στιγμή που εκατομμύρια άνθρωποι ε, μαζί με αυτούς έχουν τα βλέμματα τους τραμμένα σε εμά, πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος κύριος Ρίτσαρντ Ashworth από τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Με την ευκαιρία αυτή να μιλήσω εκ μέρους της κυβέρνησης αυτής της μεγαλειότητας θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Φερχόφστατ, ο οποίος όπως πάντα δεν κατάλαβε ακριβώς το θέμα και όπως πάντα στρέφεται προς την ε, λάθος κατεύθυνση. Αν είχε διαβάσει την έκθεση θα διαπίστωνε ότι η κυβέρνησή μας αναφέρεται ότι πρόκειται για μια περίοδο κρίσης για την Ευρώπη και ότι οι οικονομίες ε, είναι στα στασιμότητα, χάνονται θέσεις εργασίας και οι οικονομίες μας προσπαθούν να ανταγωνιστούν σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι ένας προπολογισμό που θα είναι σχετικός, που θα προσθέτει αξία και θα έχει σχέση, επαφή με τον κόσμο. Αλλά αυτό που προσφέρουν κύριο Φερχόφτατ και η συναδελφοί του είναι μία από τα ίδια. Δηλαδή, λέμε αν δεν αλλάξεις κατεύθυνση θα καταλήξεις στο σημείο για το οποίο ξεκίνησες. Εδώ χρειαζόμαστε αλλαγή κατεύθυνσης εμείς και η κυβέρνηση αυτής μεγαλειότητας. Συμφωνούμε ότι πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες του τομείς που αυξάνουν, που προσφέρουν προστιθέμενη αξία. Συμφωνούμε για την έρευνα και ανάπτυξη, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, την ενέργεια, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. Συμφωνούμε. Η παιδεία, περισσότερες επιχειρήσεις, ενθάρρυνση της ενιαίας αγοράς. Είναι σόφρονες και υγιείς επενδύσεις που θα βοηθήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης. Αυτό που δεν συμφωνούμε είναι να θεωρήσει το σώμα μας για το λόγο αυτό δικαιολογημένη το αίτημα για αυξανόμενο, αυξαμένο προπολογισμό. Ε, Σε ολόκληρη την Ευρώπη οι κυβερνήσεις επιβάλλουν προπολογισμού λιτότητας. Εδώ το σώμα μας δεν θα ήταν σωστό εάν ζητούσε το αντίθετο εάν επέλεγε να αγνοήσει την επιστολή των πέντε αρχηγών ε, κυβερνήσεων γιατί αυτό που λένε αυτοί είναι ότι η περισσότερη Ευρώπη δεν αποτελεί απάντηση. Η πιο έξυπνη Ευρώπη είναι η απάντηση. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν προπολογισμό που να στρέφεται πιο συγκεκριμένα στα διάφορα θέματα. Στην Επιτροπή Σούρε συζητήσαμε τις προτεραιότητες αλλά δεν κάναμε τίποτα επ' αυτών. Δεν υπήρχε ένδειξη, η προθυμία ότι μπορούμε να κάνουμε δύσκολες επιλογές, να αυτά που κάνουν οι διάφορες κυβερνήσεις της Ευρώπης αυτή τη στιγμή δηλαδή. Δεχόμαστε λοιπόν ότι πρέπει ότι πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες για τις νέες προτεραιότητες. Αλλά θεωρούμε επίση ότι έφτασε η στιγμή να επανεξετάσουμε τις παραδοσιακές προτεραιότητες. Και πάλι λοιπόν μια χαμένη ευκαιρία για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ε, και σας ερωτώ, θέλετε να απαντήσετε στην ερώτηση μπλε κάρτας. Συμφωνείτε, πολύ ωραία. Ο κύριος Νταφ έχει το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφό μου το εξής. Δέχεστε να μεταφερθούν βασικά στοιχεία δαπανών από εθνικούς σε ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και εάν συμβεί αυτό θα έχουμε εξοικονόμηση κόστους και οικονομίες κλίμακος. Δέχεστε ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε πράγματι να εξοικονομήσουμε χρήματα από τα Υπουργεία Οικονομικών των κρατών μελών. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνοντας ε, τη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών προοπτικών. Πρόκειται για ένα λογικό επιχείρημα το οποίο νομίζω ότι απαιτεί και μία λογική απάντηση από το Λονδίνο. Πρόεδρε, κατανοώ την ερώτηση και όπως πάντα ε, σωστά όλα στη θεωρία, στην πρακτική όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Για δείξτε μου αποδείξεις όπου μια τέτοια μεταφορά θα επέφερε ε, μεγαλύτερη εξοικονόμηση δαπανών. Για δείξτε μου πού ακριβώς εξοικονομήθηκαν χρήματα των πολιτών αντί να αυξηθούν οι δαπάνες. Αυτός ο προϋπολογισμός ε, ε, ζητάει περισσότερη Ευρώπη, αλλά όχι ευφιέστερη Ευρώπη. Η κυβέρνηση του ε, Ηνωμένου Βασιλείου ζητάει πιο σωστή χρήση των κονδυλίων και όχι αύξηση των κονδυλίων. Εκ των πρασίνων, ο ε, κύριος Άικχουτ Μπάς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το να διαπιστώνει κανεί ότι όταν πρόκειται για έναν προπολογισμό που αφορά στο μέλλον, εκείνο που συζητάμε είναι το πόσο το ύψο των κονδυλίων. Όμω θα έπρεπε να μιλήσουμε για τρία θέματα που είναι καθοριστική σημασία για του πράσινου. Πρώτον, ε, χρειαζόμαστε ένα όραμα για την Ευρώπη. Ποια είναι η υπεραξία αυτού του προγράμματο ε, σε σχέση με το, την υπεραξία. Πράγματι, ο προπολογισμό πρέπει να είναι πιο πράσινο, να είναι στραμμένο στο μέλλον. Τούτο όμω σημαίνει και μία μετατόπιση και σημαίνει χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Η τρίτη προτεραιότητα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ίδιου πόρου. Γιατί με τον τρόπο αυτό το σύστημα θα είναι περισσότερο διαφανέ και περισσότερο δίκαιο. Και για να γίνει αυτό, επαναλαμβάνω, χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδιου πόρου. Α δούμε τι τρει προτεραιότητε. Πρώτα την υπεραξία. Συζητείτε το ότι εφόσον μεταφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χάνονται σε μία μαύρη τρύπα. Μα είναι ανόητο αυτό. Είναι απόλυτα ανόητο. Για δέστε τι μπορεί να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι γιατί τα κονδύλια πρέπει να δαπανώνται σε ευρωπαϊκό και όχι σε εθνικό επίπεδο. Α δούμε την διπλωματική υπηρεσία, ε, τι πρεσβείε στο εξωτερικό. Έχουμε 27 πρεσβείε και στι χώρε Αφρική. Αυτό θέλουμε ή να έχουμε μία και μόνο πρεσβεία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αυτό θα σήμαινε ότι εξοικονομούνται χρήματα σε 27 κράτη-μέλη ας πάμε στις υποδομές. Αν ως ε, κράτη επιθυμούμε ή όταν ε, δημιουργούμε υποδομές, ε, πώς μεριμνάμε στο να υπάρχει διασυριακή σύνδεση, παραδείγματο χάνει στα ενεργειακά δίκτυα. Εκεί χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά κονδύλια ή στην καινοτομία και στην έρευνα. Πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε οικονομίες κλίμακας. Αυτό λοιπόν είναι το όραμα του μέλλοντος, αυτή είναι η ευρωπαϊκή υπεραξία και τούτο πρέπει να περιλαμβάνει ο ευρωπαϊκός προπλαγισμός. Πάμε τώρα τώρα στον προπολογισμό που είναι στραμμένος προς το μέλλον. Ο σημερινός προπολογισμός είναι αυτό που στα αγγλικά πολύ απλά λέμε business as usual, κάτι το πολύ συνηθισμένο. Θέλουμε όμως να έχουμε μια ευφυή οικονομία, μια βιώσιμη οικονομία. Σε αυτήν πρέπει να επενδύσουμε. Και οι, που προ... που... οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι τεράστιες. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα κενά. Μας λείπει εργατικό δυναμικό, μας λείπουν φυσικοί πόροι. Εκεί ακριβώς ε, καλούμεθα να επενδύσουμε. Ή το Γεωργικό Ταμείο. Και αυτό πρέπει πρέπει να ανανεωθεί, να γίνει πιο πράσινο. Να έχουμε δηλαδή ένα τομέα ο οποίο ε, θα συνδυάζεται θαυμάσια με του φυσικού πόρου. Τα διαρθρωτικά ταμεία. Και αυτά καλούνται να αντιμετωπίσουν τι νέε προκλήσει. Εξοικονόμηση ενέργεια, ε, τα διαρθρωτικά ταμεία που έχουν σχέση με την ενέργεια πρέπει να έχουν στόχο το 2020. Νέες λοιπόν προκλήσεις, ε, βιώσιμη οικονομία, ε, υποδομή για ενεργειακή πολιτική, εξωτερική πολιτική, αραβικέ χώρε, Για όλα αυτά χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά κονδύλια. Όπω επίση και για την καταπολέμηση τη φτώχεια μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά είναι ευρωπαϊκά καθήκοντα. Και όσον αφορά του ίδιου πόρου, Το σημερινό σύστημα έχει χρεοκοπήσει. Οι επιστροφέ προ του Βρετανού. Αυτό το θέλουν και οι Ολλανδοί και οι Δανείοι. Μα είναι ένα σύστημα που έχει αποτύχει. Το σύστημα πρέπει να γίνει πιο δίκαιο και περισσότερο διαφανέ. Και για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε ίδιου πόρου δικά μας εισοδήματα ή η φορολόγηση των επενδύσεων και εκεί μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα και αυτό πρέπει να γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τελειώντας λοιπόν θα ήθελα να φερθώ στο εξή. Εκείνα τα κράτη-μέλη τα οποία λένε ότι ε, παίρνουν περισσότερα χρήματα αλλά παράλληλα θέλουν να ε, δώσουν περισσότερα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλω να του πω το εξή. Αν θέλετε λιγότερα για πέστε μας σας παρακαλώ σε ποιες, από ποιε προτεραιότητες θα παραιτηθούμε γιατί αν θέλει κανείς λιγότερα χρήματα πρέπει να αποφασίσει περισσότερες προτεραιότητες με λιγότερα χρήματα με αυτό δεν γίνεται, είναι παράλογο. Αυτό λοιπόν είναι το ερώτημα που ε, στρέφεται προς την Βρετανική και την Ολλανδική κυβέρνηση. Ο κύριος Πίσκη από την, Ενωμένη, από την Ενωμένη Αριστερά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιγητά. Θα κατανοείτε βέβαια ότι η αριστερά θέτει πολύ ψηλέ ε, απαιτήσει ε, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό είμαστε απογοητευμένοι για το ότι το κοινωνικό στοιχείο στην έκθεσή σας δεν είναι πρώτη προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι η διατήρηση και η ανάπτυξη του κοινωνικού μοντέλου στην Ευρώπη και η προαγωγή της αρχής της ελεγγύη, ειδικά σε περίοδους ε, κρίσης και ειδικά σε περίοδους περικοπών, είναι πολύ σημαντικέ αρχές. Γιατί και τα δύο είναι πολιτιστικά επιτεύγματα τη Ευρώπη, τα οποία προέκυψαν από την ε, ολοκλήρωση, την σύμπλευση των ε, κρατών μελών. Αναφέρεται ότι υπάρχουν πάρα πολλές ε, προκλήσεις ε, και πέρα από τη στρατηγική για το 2020. Εγώ δεν πιστεύω ότι η αύξηση κατά 5% θα είναι αρκετή. Ως Κοινοβούλιο οφείλουμε να πούμε με απόλυτη σαφήνεια ότι πρέπει να προάγουμε ιδιαίτερα την κοινωνική Ευρώπη. Η Frontex, ε, αν θέλετε, μπορεί λιγάκι να περιμένει, δεν είναι και τόσο τραγικό αυτό, ε, το να καλούμε το Συμβούλιο να θέτει αρνητικές προτεραιότητες, δηλαδή να προβαίνει σε περικοπές, τούτο εγώ το κρίνω λάθος. Παράλληλα βέβαια, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι με την έκθεση αυτή η κοινοβουλευτική συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, η συζήτηση αυτή πράγματι πρέπει να δρομολογηθεί. Κυρίως η εισαγωγή του φόρου ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Επιτέλους, ε, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Γιατί εδώ δεν πρόκειται μόνο για ένα χρήσιμο στοιχείο χρηματοδότησης, αλλά πρόκειται και για μεγαλύτερη διαφάνεια για το πώς ακριβώς χρηματοδοτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως πρόκειται και για ένα σημαντικό τμήμα της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Κατά τη δική μου άποψη, εξίσου σημαντικό είναι να, καταργηθεί, να καταργηθούν οι επιστροφές προς τους Βρετανούς και η επαναδιοχέτευση μη απορροφημένων κονδυλίων στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. από ε, ελευθερίας. Ε, θα μας κατηγορήσουν ξανά ότι α, είμαστε πολύ μακριά από την πραγματικότητα ε, για, λόγω της αύξησης που ζητούμε. Ε, αυτό οφείλεται στη χρηματοδότηση της στρατηγικής 2020. 20. Από την μια μεριά ε, μας, ε, ε, ε λένε ότι αυτή θα μας βγάλει από την κρίση. Όμως ας δούμε τι έγινε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, σπαταλήθηκαν τα χρήματα των φιλολογημένων, δεν θα πρέπει να επαναληφθεί. Το ελεκτικό συνέδριο άλλωστε ε, αποκάλυψε σημαντικές παρατυπίες σε διάφορες πολιτικές που επιβαρύνουν με 2,8% τον προπολογισμό κάθε χρόνο. Και παρόλα αυτά αυτές οι περιοχές που είχαν προβεί σε αυτές τις παρατυπίες εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται. Ε, μεγάλες ε, καθυστερήσεις ε, παρατηρήθηκαν ενώ κάποια προγράμματα όπως το Γαλιλαίο που από 7,7 δισεκατομμύρια έφτασε στα 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμό τριπλασιάστηκε δηλαδή χωρίς τεχνολογική πρόοδο ε, το 4,7% του πληθυσμού ε, ασχολείται με τη διορκική πολιτική, η οποία λαμβάνει το 40% των ποσών. Η αλληλευτική πολιτική ε, απαιτεί από τους πολίτες να στέλνουν ένα δισεκατομμύριο ευρώ στις Βρυξέλλες κάθε χρόνο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικών ε, εξωτερικής δράσης Δράση κοστίζει 100 δισεκατομμύρια κάθε χρόνο και παρόλα αυτά δεν έχει δώσει αποτελέσματα. Όλα αυτά είναι παραδείγματα ε, τα οποία θα δικαιολογούσαν μείωση, όχι ε, πάγωμα του προπολογισμού, μείωση. Ε, ελπίζω ότι η Βρετανική κυβέρνηση θα στυλώσει τα πόδια της και θα πει φτάνει πια. Ε, παρόλο ότι δεν ζητά αυτή τη στιγμή μείωση αλλά μόνο πάγωμα. Ο κύριος Χάρτονγκ, εκ μέρους των μη εγγεγραμμένων. Ε, μιλούμε για τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά το 2013 ε, μιλάμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, τα επόμενα χρόνια και ε, ε ειλικρινά δεν θα πρέπει να παραδοθούμε στην δικτατορία της ελίτ σε εθνικό επίπεδο, των ελίτ σε εθνικό επίπεδο. η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα από τα κράτη-μέλη, χωρίς να αγνοεί όμως ε, την κυριαρχία ε, των ε, εθνικών των χωρών. Ε, εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να συμφωνήσουμε με αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι θα έπρεπε να πεταχτεί στα σκουπίδια. Γιατί με αυτή την έκθεση θα σβήσουμε τα φώτα στην Ευρώπη και θα προετοιμάσουμε ένα πιο σκοτεινό μέλλον για τα παιδιά μα. Εμεί θέλουμε να διατηρηθούν αναμένα τα φώτα και θα καταψηφίσουν την έκθεση. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπω βλέπετε, κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση για το μέλλον τη Ευρώπη και περιμένουμε την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Α, μπλε κάρτα. Είστε διατεθειμένος να απαντήσετε, κυρία Χαρτόγκ. Ε, ναι. Ο κύριος Γκάρτ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια ερώτηση έχω προς τον κύριο Χάρτονγκ. Αυτή τη στιγμή πολλά κράτη-μέλη είναι μέλη των G8. Εκπροσωπούνται εκεί, που είναι στον οργανισμό των 8 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Σε 10-15 χρόνια ούτε ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής ε, Ένωση δεν θα αντιπροσωπεύεται εκεί. Πώ μπορείτε να ισχυρίζεστε ότι οι διάφορε ευρωπαϊκέ χώρε θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Δεν θεωρείτε ότι η μόνη λύση είναι να προχωρήσουμε με την Ευρώπη, να είμαστε και πάλι όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Voorzitter, ik eh, bedank mijn collega voor Ευχαριστώ τον συνάδελφο για την ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Η Ευρώπη είναι καταπληκτική και δυνατή λόγω των κρατών μελών της και τα κράτη-μέλη συνεργάζονται έχουν μελετήσει τα πράγματα και πραγματικά μπορούν να έχουν μια ισχυρή φωνή στον κόσμο. Έτσι θα γίνει και στο μέλλον. Και ακριβώς επειδή συνεργάζονται καλά οι εθνικές κυβερνήσεις θα υπάρξει μια εξαιρετική φωνή της Ευρώπης στο μέλλον. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα ακούσουμε την ευρωπαϊκή, ε, άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ευπρόσδεκτη η έκθεση της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ. Είναι πραγματική συνεισφορά στην προετοιμασία των ε, επερχόμενων δημοσιονομικών προοπτικών μια πραγματική ευρωπαϊκή έκθεση, μια πραγματική ευρωπαϊκή προοπτική για το ευρωπαϊκό έργο. Είναι κάτι που το απε... απολύτως χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι έχουμε κοινά προβλήματα που απαιτούν κοινή απάντηση σε μια εποχή που όπως είπε ο κύριος Σούλτς είναι μια εποχή όπου διακυβεύεται η αλληλεγγύη. αλληλεγγύη. Όμως ε, συμμετείχα στην Επιτροπή Σούρε και έγινα, υπήρχαν ε, διαφωνίες ε, ξέρω για ποιο λόγο ήταν πολύ καλή η διαχείριση ε, της συζήτησης. Εδώ μιλάμε για ευρεία συνένεση, αλλά είχαμε πλειοψηφική ψήφο, η οποία ελπίζω ότι σήμερα θα επιβεβαιωθεί στην Ολομέλεια. Πραγματικά υπάρχει ένα όραμα στην έκθεση αυτή. Ναι, λέμε επίσης ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό δεν ε, ενδιαφέρεται να γίνει μια επανάληψη των εθνικών προϋπολογισμών αλλά θέλει να προσπαθήσει την επιδίωξη των κοινών στόχων πέρα των δυνατοτήτων των εθνικών κρατών μελών όπου μπορούμε ως Ευρώπη να κάνουμε οικονομίες κλίμακας και μεγάλες συνέργειες. Πραγματικά πρέπει να συμβεί αυτό εκεί όπου έχει μια διαφορά, που έχει νόημα εκεί που ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα κάνει σωστές επενδύσεις για την αντιμετώπιση των ε, ελλημάτων. Έχουμε τις, κοινές αγροτι... τις παραδοσιακές πολιτικές, κοινή αγροτική πολιτική και πολιτική συνοχής. Παραδοσιακές αλλά όχι ξεπερασμένες. Αλλά μιλάμε για το μηχανισμό επίτευξης των των στόχων της στρατηγικής του 2020 όταν έχουν σωστή διαμόρφωση στον προϋπολογισμό δημιουργούν περιθώριο για πολύ ουσιαστικά καλύτερη χρηματοδότηση η καινοτομία και η διαχείριση, στη διαχείριση ας πούμε των ροών μετανάστευσης και οι εξωτερικές ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι τώρα πολύ έντονες σε περιοχές όπως η Μεσόγειο. Μιλάμε για την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά μιλάμε κυρίως για το πώς θα διασυνδεθεί η Ευρώπη μέσω των διαευρωπαϊκών δίκτυων και των διαμεθοριακών συνδετικών αγωγών των ενεργειακών δικτύων. Πρέπει να αποκτήσει νέες λειτουργίες όπως ένα ε, toolbox για, την, ε, για, δημόσια, για τα δημόσια οικονομικά και ως εγγύηση για την ε, ισοσκέληση του προϋπολογισμού αλλά και για το ισοζύγιο πληρωμών αλλά και για πιο ε, καινοτόμα εργαλεία που θα μοχλεύσουν ε, τα οικονομικά. Ζητάμε μια μεταρρύθμιση, ζητείτε μια μεταρρύθμιση ε, των οικονομικών και πραγματικά, όπως είπε ο κύριος Ντόλ, έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Να διευκολύνουμε τη ζωή των Υπουργών Οικονομικών δίνοντας νέους ιδίους πόρους στον προϋπολογισμό. Το πακέτο του Ιουνίου θα υποβληθεί στο τέλος Ιουνίου μιλάει για νούμερα, ε, για το τον πολιετή κανονισμό, διαθεσμική συμφωνία και για τους ιδίους πόρους. Συγκεκριμένες κλαδικές προτάσεις θα εμφανιστούν αργότερα το, μεταξύ Σεπτεμβρίου και του τέλους του έτους. Ολοκληρώνοντας θέλω να, για μια ακόμα φορά να επαναλάβω την πεποίθησή μου ότι η έκθεση της Επιτροπής Σούρε είναι καλή συνεισφορά στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς για την Κομισιόν. Η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απαραίτητη όχι μόνο για την καλή αρχή και τη διαμόρφωση αυτής της πρότασης αλλά για την ευτυχή ολοκλήρωση των εξαιρετικά δύσκολων διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δύο θεσμικά όργανα που θέλουν να αλληλοστηρίζονται, ε, πρέπει να έχουν παρόμοια προσέγγιση στα πι και θα δείτε ότι το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υποβληθεί στο τέλος αυτού του μήνα και θα παρουσιαστεί επίσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, μπλε κάρτα. Όμως ο κανόνας αυτός δεν προβλέπεται για τους προσκεκλημένους ομιλητές. Λυπάμαι. Απευθύνεται στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εντάξει. Οπότε, περνάμε στις επιτροπές. Επιτροπή Ανάπτυξης, ο, ο συνάδελφος ε, της Μπέρμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης, ε, εδώ έχουμε να κάνουμε με μία καθοριστική σημασίας έκθεση γιατί ορίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τις ευθύνες που φέρει απέναντι ε, στα αναπτυσσόμενα κράτη ε, και κατόπιν τούτου το 0,7% του ΑΕΠ ε, που αναφέρεται εδώ αυτό δεν μας ικανοποιεί. Στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμούμε να αποφύγουμε επικαλύψεις και να γίνουμε αποτελεσματικότεροι. Ε, θέλουμε να ληφθούν μέτρα ε, που να αντιμετωπίζουν την κλιματική αλλαγή. Αυτά όμως πρέπει να χρηματοδοτούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κονδύλια όμως ε, χρειάζονται και τα κράτη-μέλη. Πέρα από τις επιδοτήσεις, τα ανθρωπιστικής φύσεως μέτρα, αυτά ε, χρειάζονται το δικό τους ε, χρηματοδοτικό εργαλείο, γιατί τα μέτρα αυτά θα πρέπει να δείχνουν και το πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα έξω. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να είναι ο σημαντικότερος εταίρος των αναπτυσσομένων κρατών και αυτό νομίζω ότι θα παραμείνει έτσι και στο μέλλον. Ε, ο επόμενος ομιλητής είναι ο Γκέρμπεν Γιάν Γκερμπράντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι ικανοποιημένη από την έκθεση ως έχει. Δίνεται έμφαση στην έλλειψη των φυσικών πόρων, μελετά την βιοπικιλότητα, την βιωσιμότητα και, αυτό που είναι σημαντικό, αναγνωρίζει την σημασία της βιωσιμότητα για τις οικονομίες μα. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή κάθε κράτος μέλος προσπαθεί να μετρήσει κάθε δεκάρα πριν την δαπανίσει και κάνουμε κάτι περίεργο. Ξοδεύουμε εκατομμύρια σε επιδοτήσεις για τομείς όπου πρέπει να μελετήσουμε καλύτερα. Η ομάδα μου υπέβαλε μια τροπολογία η οποία δεν εγκρίθηκε. Και έτσι από τώρα μέχρι το 2020 οι επιδοτήσεις οι οποίες βλάπτουν το περιβάλλον θα πρέπει να καταργηθούν. Κυρίως επειδή ζούμε σε περίοδο ελήψεων δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοιου είδους επιδοτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής από την ΕΜΒΗ περνάμε στην κυρία Κρέιλ της Περιφερειακής Ανάπτυξης γιατί οι ε, Επιτροπές Ήτρε και Μεταφορών δεν παρίστανται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική συνοχή ε, είναι ε, ένας από τους μεγαλύτερους μεμονωμένους προϋπολογισμούς Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι πρέπει να έχουμε μια νέα πολιτική που θα είναι προσαρμοσμένη και στις νέες προκλήσεις. Επιθυμούμε λοιπόν να επενδύσουμε στις επενδύσεις, επενδύσεις στην έρευνα, την καινοτομία, την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Επιθυμούμε να υπάρχει μια βιώσιμη ανάπτυξη και θέλουμε να έχουμε και τους ε, ε, εργαζόμενους με τα απαραίτητα προσόντα. Χρειαζόμαστε λοιπόν την στήριξη των περιφερειών για να καταστούν αυτές ανταγωνιστικές και να αναπτύξουν τις οικονομίες τους. Παράλληλα όμως πρέπει να πούμε ότι όλες οι περιφέρειες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην πολιτική συνοχή. Αυτό ισχύει και για τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης ε, και Ανατολική Γερμανία χρειάζεται στήριξη. Βέβαια όχι μόνο αυτή και η Δυτική Γερμανία ακριβώς όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να γίνουν όλα αυτά χρειαζόμαστε ένα προπολογισμό που δεν μπορεί να είναι μικρότερος ε, του τρέχοντος και δεν μπορεί να είναι και κατακαιρματισμένο σε διάφορους τομείς. Οφείλουμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια και όλα αυτά να τα συνδυάσουμε με την κατάργηση της περιττής γραφειοκρατίας. Η συνοχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλληλεγγύη, όμως η συνοχή είναι και λογικά και οικονομικά λογική. Ε, κατόπιν τούτου ας προσπαθήσουμε λοιπόν την ε, χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής να την θεωρήσουμε προτεραιότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή για το ότι έλαβε υπόψη του τη θέση της ε, Επιτροπής ε, Περιφερειών, της Περιφερειακής Επιτροπής και επίσης θα ήθελα να πω ότι πράγματι πρέπει να βελτιωθούν και ενδιάμεσε κατηγορίες. Στην Επιτροπή Περιφερειών καταλήξαμε σε ένα συμβασμό και επιθυμώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τον συμβασμό αυτό, οποίο εκφράζουμε εμείς μέσα από την έκθεση Γκαρίγκα. Και για το λόγο αυτό ε, ζητούμε την σύμφωνη γνώμη σας. Ο συνάδελφος κύριος Τζοβάνι Λαβία από την Επιτροπή Γεωργίας. Κύριε Πρόεδρε, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και εγώ εκ μέρου ε, των ε, περισσότερων συναδέλφων της Επιτροπής Γεωργίας να συγχαρώ τον συνάδελφο, τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε τους τελευταίους μήνες. Η συζήτηση για τις δημοσιονομικές προοπτικές ήταν πολύ έντονη τελικά προέκυψε μια σύνθεση απόψεων η οποία παρουσιάζει τις ε, θέσεις των διαφόρων εθνικών αντιπροσωπείων και των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Επειδή είμαι εισηγητής ε, γνωμοδότησης ε, της Επιτροπής Γεωργίας πρέπει να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με το ότι πρέπει να παραμείνει απαράλλαχτος ο δικός μας ο γεωργικός προϋπολογισμός. Και όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι από την ίδια Επιτροπή είμαι κατά της τροπολογίας της Επιτροπής των Φιλελευθέρων που επιθυμούν να περικοπούν τα κονδύλια που δίνουν τη Γεωργία για να χρηματοδοτηθούν άλλε προτεραιότητε. Μην ξεχνάτε, συνάδελφοι, ότι η κοινή γεωργική πολιτική προβλέπεται από τι συνθήκε και είναι μία από τι λίγε ουσιαστικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε ένα στρατηγικό τομέα γιατί προσφέρει ένα, μια αυθεντική ευρωπαϊκή υπεραξία. Ευχαριστώ. Κυρία Σόριν Καταλήν σοριν καταλιν ιβαν ο, ναι, ο κύριος. Ε, όταν μιλάμε για ε, το επόμενο πι πι, μιλούμε ασφαλώς και για την ευρωπαϊκή υπεραξία. Και η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία ε, ε αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο στον δικό μου τομέα ε, διότι ο πολιτισμός και είναι η πραγματικό μας ατού και οι νέοι θα πρέπει να ε, κατανοήσουν την αξία της Ευρώπης. Ε, τα σχέδια για τους νέους, τα σχέδια για την παιδεία και την εκπαίδευση θα πρέπει να έχουν αυξημένο προπολογισμό στο μέλλον. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό και στην ε, νεότητα στο μέλλον. Είναι προτεραιότητά μας, όπως και ο αθλητισμός. Ευχαριστώ. Η κυρία Σβένσον από την ε, Επιτροπή για Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Πρόβλημα. Πρόβλημα με το μικρόφωνο. Εντάξει, ωραία. Εγώ συνέταξα την δική μας ε, γνωμοδότηση στην Επιτροπή μας και θέλω να πω ότι μιλούμε για μια σημαντική απόφαση, μιλούμε για οικονομικά θέματα που έχουν σχέση με την δημοσιονομική πολιτική, την εμπορική πολιτική κλπ. Ζητήματα τα οποία ε, επηρεάζουν άμεσα τον προπολογισμό. Αυτό που βλέπουμε όμως ε, είναι ότι δεν γίνεται πολλής λόγος για άλλα ζητήματα. Αν θέλουμε σύγχρονο Προπολογισμό θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα σημαντικά θέματα για το μέλλον και να τα συμπεριλάβουμε ήδη από σήμερα στον προπολογισμό. Τα προσόντα των γυναικών, για παράδειγμα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η εμπειρία τους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Χρειαζόμαστε ε, κατάρτιση προπολογισμού με βάση το φύλλο, λαμβάνοντα υπόψη το φύλλο. Μιλούμε για αύξηση του προπολογισμού, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Χρειαζόμαστε και την ε, πολιτική γενναιότητα ε, να ε, αντικατοπτρίσουμε τις προτεραιότητες μας στην ίδια μας την εργασία, στην ίδια μας τη δουλειά. Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη και να χρησιμοποιήσουμε τα προσόντα και την εμπειρία των γυναικών. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε πιο αποτελεσματικά τον προπολογισμό που διαθέτουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση που έχει κατατεθεί είναι μια πολύ καλή προσφορά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την ε, αντιμετώπιση της κρίσης. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον εισηγητή, τον κύριο Γκαρίγκα και την κυρία Γιούτα Χάουκ, ε, γιατί και οι δύο εργάστηκαν πραγματικά με εντυπωσιακό τρόπο εμείς ως πολιτικές ομάδες σαφώς και έχουμε διαφορές, όμως η δουλειά μας όλων μας ήταν να αναζητήσουμε ευρωπαϊκές λύσεις. Και νομίζω ότι αυτό το πνεύμα που διέπνευσε μας θα μπορούσε να διαπνεύσει και άλλα όργανα. Πέρα λοιπόν από περαιτέρω έσοδα, ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους. Εμείς λοιπόν θα παραμείνουμε ε, πιστοί στις συνθήκες αν ε, συνεχίσουμε αυτό αυτό ε, και στο μέλλον και δεν πρέπει πλέον να υπάρχουν επιστροφές. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το σεβαστούν πάρα πολλές πρωτεύουσε και θα πρέπει να το συζητήσουν και με τους αδέλφους του στα Εθνικά Κοινοβούλια. Εμείς θέλουμε να διαφυλάξουμε την ενότητα του προεπολογισμού και οι διάφορες πολιτικές να μην ε, βγουν από τον ευρωπαϊκό προεπολογισμό. Όταν μιλάμε λοιπόν για καθήκοντα, μιλάμε κατ' ουσίαν για τις υποχρεώσεις που πορεύουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουμε τη στρατηγική του 2020 όλοι δεσμευτήκαμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη στρατηγική ανάπτυξη ως βάση για την κοινωνική δράση και μέσα από την ευρωπαϊκή υπεραξία και τη συζήτηση για την απαραίτητη συνέργεια που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους εθνικούς και τον ευρωπαϊκό προπλογισμό μέσα από όλα αυτά πρέπει να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε τις συζητήσεις ανεξάρτητα βέβαια από τις περικοπές που υπάρχουν στον ευρωπαϊκό προπλογισμό μπορούμε θεωρώ πράγματι να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τη σχέση και τη συνέργεια, αν θέλετε, ανάμεσα σε εθνικού και ευρωπαϊκό προβλησμό. Στο Συμβούλιο πρέπει να είναι σαφέ ότι αν δεν συνεχιστεί αυτό ο δρόμο, τότε το Συμβούλιο πρέπει να μα πει ποιε είναι οι δικέ του πολιτικέ προτεραιότητε, ποιε θα διαγράψει, ποιε θα πάψει να χρηματοδοτεί. Αυτή είναι μια αλήθεια που πρέπει να αναφέρουμε στου πολίτε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιδράσει θετικά στι προτάσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εγώ προσβλέπω στο ότι οι επόμενε προεδρίε θα βρουν ένα δρόμο για να συζητήσουν καθαρά και ειλικρινά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κοιτάξτε, αν θέλετε ε, μπορείτε να μιλήσετε και για άλλο ένα λεπτό γιατί σας έχει υποπληθεί η διαδικασία της μπλε κάρτας. Το δέχεστε? Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Κοιτάξτε, εξ όσων γνωρίζω, ο συνάδελφο κύριος Μπέγκε είναι μέλος ε, των χριστιανοδημοκρατών στην Γερμανία και διαρωτώ με ε, αυτά που μας είπε είναι η προσωπική του θέση ή είναι η θέση των χριστιανοδημοκρατών στη Γερμανία. Συνάδελφε. Ε, πολύ ευχαρίστω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Πράγματι, εγώ όχι μόνο είμαι μέλο των Χριστιανοδημοκρατών, αλλά εδώ και 13 χρόνια είμαι και αντιπρόεδρο των Χριστιανοδημοκρατών στο κρατήδιο του Schleswig Holstein. Έχουμε λοιπόν μία θέση εμεί ω Χριστιανοδημοκράτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση τα οποία καταλήγουμε στο ότι οι διπόροι, πόροι, του οποίου οι αποφάσισαν, ενέκριναν οι ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η δική μας η θέση. Αλλά μπορεί να είναι σε αντίφαση με τη θέση των δημοκρατών στη Γερμανία, όμως είναι σε απόλυτη ταύτιση με την άποψη της Επιτροπής Σούρε, στην οποία ήμουνα μέλος και γι' αυτό παραμένω πιστός στα καθήκοντά μου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ε, αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις ε, για το μέλλον. Θα πρέπει να λήξει η οικονομική κρίση και να αποφύγουμε μελλοντικέ κρίσεις. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας στο μέλλον, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Χρειαζόμαστε σημαντικές διασυνορικές ε, επενδύσεις, για παράδειγμα σε θέματα όπως η έρευνα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε προβλήματα περιβαλλοντικά, κλιματικών αλλαγών, παρκούς τροφοδοσίας, ενεργειακής τροφοδοσίας. Θα πρέπει να αποφύγουμε την ε, μονιμοποίηση, ε, την, ε, την αύξηση της ανεργίας σε μόνιμη βάση. Αυτό όμως που περισσότερο χρειαζόμαστε είναι αλληλεγγύη, μια Ευρώπη να λειτουργεί πραγματικά, σωστά. Δυστυχώς όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν απειλές ακόμα και στην ίδια την ένα της Ευρώπης. Για παράδειγμα, σε αυτή την συζήτηση για τον περιπολισμό στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ, Έγινε αντιληπτό ότι πολλά κράτη-μέλη κάνουν περικοπές στον εθνικό τους προπολογισμό και φαίνεται λίγο παράξενο εμεί να ζητάμε περισσότερα χρήματα για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Όμως ταυτόχρονα θα ήταν παράλογο να αμελείς να, ε, να αγνοήσουμε τις προκλήσεις που μας περιμένουν ε, και να υποχωρήσουμε εναντί των φιλοδόξων ε, σχεδίων τα οποία έχουν αναθέσει στην Ευρώπη τα ίδια τα κράτη-μέλη πρέπει να δούμε την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία ε, και να τις βοηθήσουμε. Αν όμως μειωθεί ο προπολογισμό, δεν θα μπορέσουμε να τους δώσουμε τη βοήθεια που χρειάζονται. Η Βρετανική κυβέρνηση μιλάει για συνσφέροντες στον, ε, στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ναι, εντάξει, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία, ε, διότι θα πρέπει να δούμε τις παραδοσιακές πολιτικές και να τις ισορροπήσουμε με τις καινούριες προτεραιότητες μας. Ζητούμε 5% αύξηση και συγχαίρω τον κύριο Γκάρικα που εξασφάλισε σημαντική υποστήριξη της πλειοψηφίας σε αυτή την έκθεση. Αυτό το 5% θα πρέπει όμως να ε, δαπανηθεί σε επενδύσεις για βασικτομής τομείς κλειδιά για το μέλλον. Για παράδειγμα, ανάπτυξη, απασχόληση, έρευνα. Όλα αυτά χρειάζονται χρήματα. Και χωρίς την κατάλληλη χρηματοδότηση δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Επίσης, θα πρέπει να αλλάξουμε προσέγγιση. Ε, ε, η Σουηδία μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη δεκαετία του 1990 και ο ευρωπαϊκός προπολογισμό αυξήθηκε πιο αργά από ότι αυξήθηκαν οι εθνικοί προπολογισμοί από τότε. Για παράδειγμα, ο Βρετανικός προπολογισμό κάτι που η αυτής μεγαλειότητα δεν το αναφέρει, ε, έχει αυξηθεί περισσότερο από ότι ο ευρωπαϊκός προπολογισμό όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, θα πρέπει, να ε, χρειάζεται δημοσιονομική πειθαρχία, χρειάζεται λιτότητα, αλλά χρειάζονται και επενδύσεις για να βγούμε από την κρίση. ε, ο συνάδελφος Καρλ Χάγκλουντ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον εισηγητή για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Συγκέντρωσε όλες τις ιδέες που εκφράζονται εδώ. Γιατί οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι σοβαρές. Πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν αρκετά χρήματα και πρέπει να πετύχουμε μια ισορροπία. Εντός της Επιτροπής συζητήσαμε για αύξηση του προπολογισμού στο μέλλον κατά 5%. Ίσως το 5% να ακούγεται πολύ. Ιδίω αν πρέπει κανεί να γυρίσει πίσω στην πατρίδα του και να τα δικαιολογήσει. Αυτά όμω χρειάζονται για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στι προκλήσει του μέλλοντο και τα νέα έργα τα οποία πρέπει να φέρουμε. Χωρί χρήματα αυτό δεν θα το πετύχουμε. Πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι και για να μπορούμε να πάρουμε όλο και περισσότερα χρήματα θα πρέπει να επανεξετάσουμε το κόστος και τις υφιστάμενες δομές και να κάνουμε οικονομίες, να ε, αλλάξουμε τις προτεραιότητες εντός του προϋπολογισμού. Σχετικά έχω κατά νου την κοινή αγροτική πολιτική παραδείγματο χάρη. Επίσης την πολιτική συνοχής, γιατί μερικές φορές δεν είναι τόσο μεγάλη επιτυχία τους όσο θα θέλαμε. Συζητάμε για πολλή γραφειοκρατία το Στρασβούργο, ας πούμε, είναι ένα άλλο παράδειγμα. Εντός της ομάδα μας είπαμε πολλές περιπτώσεις που θα μπορούσε να συζητηθούν για να ζητήσουμε, να είμαστε πιο αξιόπιστοι όταν ζητάμε περισσότερα χρήματα. Είμαστε υπέρ της έκθεσης. Όχι όμως 100%. Θα ζητάμε λοιπόν μερικές φορές να θα πατήσουμε το κόκκινο κουμπί μερικές φορές και άλλες φορές το άλλο κουμπί. Όμως Πρέπει να επιδιώξουμε νέους πόρους, αλλά πρέπει να δούμε και πώς δαπανούμε τους υφιστάμενους. Η ομάδα μας είναι ξεκάθαρη, η Επιτροπή μας είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μα. Ναι, οι πόροι είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να δούμε τα προβλήματα των υφιστάμενων χρηματοδοτικών δομών. Μιλάμε για επιστροφές, ασαφεί ρυθμίσει. Δεν μπορούν αυτά να συνεχιστούν στο μέλλον. Πρέπει να προχωρήσουμε σε επικοδομητικό διάλογο με το Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό του αξιόπιστου ε, ε, προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριο Σιμάνσκι. Ε, η, η έκθεση αυτή για τα πι δέλτα πι ε, δεν σημαίνει ότι επειδή υποστηρίζεται από μας δεν έχει και αδυναμίες. Ε, χάνουμε χρόνο σε πολλά πράγματα θέλουμε περισσότερους, ζητάμε περισσότερους φόρους και οι Ευρωπαίοι έχουν ήδη να πληρώσουν πάρα πολλούς φόρους και εισφορές. Πρέπει να κοιτάξουμε με κριτικό μάτι τις πολιτικές μας και να μην αγνοούμε κάποιες σπατάλες που κάνουμε. Γιατί αν το συνεχίσουμε αυτό θα είμαστε ανέντιμοι. Στα πλαίσια της Ατζέντα 2020, μάλλον η Ατζέντα του 2020 έχει γίνει ένας γενικός στόχος. Αυτό όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε βάρος της πολιτικής συνοχής. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία η οποία ακριβώς εκεί βρίσκεται. Ένα καλό παράδειγμα εδώ είναι η Πολωνία. Βλέπουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής. Προκαλεί ανάπτυξη και αυτό ωφελεί όχι μόνο την Πολωνία αλλά συνολικά την Ευρώπη. Έτσι έχουμε περισσότερες επενδύσεις και ωφέλη όχι μόνο στη Βαρσοβία και την Πράγα αλλά και στο Άμστερνταμ, το Βερολίνο ή το Λονδίνο. Ευχαριστώ η κυρία Χέλγα Τρούπερ. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, εγώ ξεκινάω ε, με, αναφέρομαι σε αυτά που είπε ο κ. ο οποίο ζήτησε έναν ευφιέστερο ευρωπαϊκό πολιτισμό και λέει ότι αυτό είναι καλύτερο από έναν υψηλό ευρωπαϊκό προπολογισμό. Λάθο το δίλημα. Πρέπει να έχουμε σωστή, έξυπνη ευρωπαϊκή πολιτική, παράλληλα όμω να εντοπίσουμε πού μπορούμε να κάνουμε περικοπέ, καλύτερη διαχείριση, ε, πού μπορούμε να συγκρατήσουμε τι δαπάνε. Αυτή η ειδική λοιπόν επιτροπή, η ΣΟΥΡΕ, είχε ως καθήκον να εντοπίσει ε, πόσα κονδύλια ακριβώ ε, χρειαζόμαστε έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Πρόκειται δηλαδή για μεταρρυθμίσεις, για πολιτικό θάρρος και επίση εκείνο που ενδιαφέρει είναι να έχουμε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις μεγάλες προκλήσεις μέχρι το 2020. Με τη δική σας την απάντηση κύριε Ashworth ε, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Ο κύριος Μπέγκε πολύ σωστά μίλησε. Κατά την άποψή μου πιστό στις συνθήκες λέει ναι πρέπει να έχουμε το θάρρος να επανέλθουμε σε ένα σύστημα των αυθεντικών ίδιων πόρων. Αυτό κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο δυνατή. Το σύστημα το δικό μας της χρηματοδότησης καθίσταται διαφανέστερο. Οι πολίτες γνωρίζουν από πού προέρχονται τα χρήματα και ως πράσινοι θέλω να σας πω ότι εμείς έχουμε ιδιαίτερα κατά νου τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών γιατί ο φόρος αυτός θα ρυθμίσει τις αγορές και θα μας προσφέρει τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε μια πιο έξυπνη πολιτική. Αυτό είναι ο δρόμος προς το μέλλον που δεν θα στραγγαλίσει τα κράτη-μέλη αλλά θα δώσει σε όλους μας νέες προοπτικές. Γι' αυτό λοιπόν και ο κύριος Φερχόφ στατ έχει δίκιο, που λέει βεβαίω και πρέπει να είμαστε έτοιμοι στην περίπτωση αυτή να αντιμετωπίσουμε κοινά ευρωπαϊκά καθήκοντα. Να έχουμε ευρωπαϊκή διπλωματική υπηρεσία και παράλληλα να κάνουμε και εθνικέ περικοπέ. Όχι το ένα ει βάρο του άλλου. Όχι. Ευρωπαϊκή ευθύνη σημαίνει ότι περιορίζει κανεί τι εθνικέ αρμοδιότητε και τι μεταθέτει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξέρετε γιατί. Γιατί θέλουμε να είμαστε πιο ισχυροί. Θέλουμε την ευρωπαϊκή υπεραξία που είναι καλή για τον πολίτη στην πολιτική έρευνα στην εκπαιδευτική πολιτική. Αυτά είναι τα μεγάλα καθήκοντα που μας περιμένουν. Η οικολογική μεταρρύθμιση, να συστήσουμε ευφυή ενεργειακά δίκτυα. Ε, χρειαζόμαστε χρήματα όπως και για τις ευρυζωνικές διασυνδέσεις. Ε, για όλα αυτά λοιπόν χρειαζόμαστε έναν έξυπνο και έναν λογικό προϋπολογισμό. Μπορείτε, δέχεστε μία μπλε κάρτα, θα απαντήσετε σε μπλε κάρτα. Συνάδελφος ε, Βαν Ντάλεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Τρούπελ, Η κυρία Τρούπελ προβαίνει στις ίδιες ε, μεγαλοστομίες, περισσότερη Ευρώπη, καλή Ευρώπη και περισσότερη Ευρώπη σημαίνει περισσότερα χρήματα. Γνωρίζουμε όμως ε, τα ποσοστά ε, τα οποία επιθυμείτε εσείς και ο κύριος Φερχόφτσατ. Αν όμως όλα αυτά ισχύουν κυρία Τρούπελ, τότε είναι πολύ περίεργο ότι οι πολίτες βλέπουν τα πράγματα διαφορετικά. Ε, μειώνεται η εμπιστοσύνη τους προς την Ευρώπη και οι πολίτες βλέπουν την Ευρώπη ως μια κρέατομηχανή που απορροφά όλο και περισσότερα κονδύλια. Μήπως θα ήταν καιρός κυρία Τρούπελ να αλλάξετε λιγάκι τις απόψεις και να πάτε προ την κατεύθυνση του κυρίου Ashworth. Η κυρία Τρούπελ, συνάδελφε, νομίζω ότι εδώ κάνετε ένα τραγικό πολιτικό λάθος. Ε, εάν ε, στην Ευρώπη όπιστο δρομήσουμε πίσω στα εθνικά στα κράτη-μέλη, τότε θα καταστρέψουμε ε, τα τελευταία 15 χρόνια όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Και τι θα κάνουμε, θα αγνοήσουμε τη δωροδοκία Εκεί πράγματι πρέπει να επέμβουμε, εκεί συμφωνώ μαζί σας, όμως αυτό που ενδιαφέρει είναι να συνεχίσουμε να παράγουμε ευρωπαϊκή υπεραξία. Τα εθνικά κράτη μόνα τους ε, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον διεθνή ανταγωνισμό. Τα κράτη-μέλη μόνα τους, 27, δεν μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Μόνο λοιπόν αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας θα καταφέρουμε κάτι. Αυτό το κάναμε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσουμε και όχι να φαλκιδεύσουμε τις προσπάθειες. Ο κ. Πόρτας. Ακούω εδώ και ώρα αυτή τη συζήτηση και, παρόλα, και η δική μου άποψη είναι λίγο αιρετική. Η ερώτηση είναι εξή. Είναι βιώσιμο ένα νόμισμα χωρίς ισχυρό ευρωπαϊκό προπολογισμό. Η δική μου απάντηση είναι όχι. Αυτό δεν είναι δυνατόν και η κρίση δημοσίου χρέου ακριβώς αυτό αποδεικνύει. Αποδεικνύει ότι αν σήμερα είχαμε ένα ισχυρό προπολογισμό, δεν θα ήταν δυνατές κερδοσκοπικές επιθέσεις εναντίον του δημόσιου χρέους της Ελλάδας ή της Πορτογαλίας. Και σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Ε, στο, το βασικό ερώτημα στο οποίο δεν απαντάει η έκθεση. Λείπει φιλοδοξία η οριακή αύξηση του 5% στον προπολογισμό φαίνεται πολύ, ε, ακόμα και αυτή φαίνεται πολύ στη, στα μάτια της, ε, της μεγαλειότητας ε, της κυβέρνησης της Βρετανίας. Όμως, είναι αρκετό αυτό το μικρό ποσοστό είναι αρκετό το πάγωμα που προτείνουν πολλοί για να ανταποκριθούμε στις καινούργιε δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει με την καινούργια συνθήκη, στις προτεραιότητές μας για το μέλλον. Η πολιτική συνοχής μπορεί να εξακολουθήσει να ισχύει όταν αρχίζουμε, αρχίζουμε να ε, ε, επιστρέφουμε στην παλιά κατάσταση. Εμείς θα υπερψηφίσουμε την έκθεση. Αλλά διακόπτει ο πρόεδρος τον ομιλητή. Η κυρία Τζαβέλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούστηκαν πολλά και θέλω και εγώ, εγώ να μιλήσω διαφορετικά. Πριν από κάποια χρόνια έτρωγα με τον αείμνηστο πρόεδρο Τζέραλ Ford των Ηνωμένων Πολιτειών και μου υπε... περιέγραφε πώς φτιάχτηκε η ομάδα των G7. Είπε ότι ήθελε να συναντηθεί με τον Κάλαχαν, αν δεν απατώ, με τον τότε πρωθυπουργό της Βρετανίας, για κάποια ζητήματα. Και ο Κάλαχαν είπε, γιατί να μην το συνδυάσουμε με ένα ωραίο παιχνίδι γκολφ. Και είπε ο Φόρντ. Και ο Τριντό, ο, πρόεδρο, Πρωθυπουργό του Καναδά παίζει καλά, να τον καλέσουμε και αυτόν. Και είπε ο Τριντό ε, που δέχτηκε την πρόσκληση. Θέλω κάποια ζητήματα που με απασχολούν, έχω κάποια ζητήματα που με απασχολούν με τους Γάλλους, γιατί δεν καλούμε και τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας. Όταν όμως το συζήτησαν τηλεφωνικά είπαν «Α, δεν θα αρέσει αυτό στους Γερμανούς, τι να κάνουμε, πρέπει να τους καλέσουμε και αυτούς». Και όταν δέχτηκαν την πρόσκληση οι Γερμανοί είπαν η Ιταλία προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμεινο, πρέπει να παρίσταται. Και μου είπε ο Φόρτ, ξέρεις Νίκη, ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι έχετε Ένωση που είναι τόσο διαιρεμένη και πάρα, χωρίς καμία ισορροπία. Κάποια στιγμή πρέπει να έχετε έναν αρκετά ισχυρό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να μπορέσετε να ανταγωνιστείτε παγκοσμίω. Ο κόσμος είναι σκληρός, πρέπει να προσέχετε. Κύριε Πρόεδρε, ως Ευρωβουλευτής ε, χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Αγγέλικα Βέρτμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Επιτροπή Προπολογισμών εδώ και μεγάλο αρκετό και αρκετό καιρό ασχολείται με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η εισήγηση του συναδέλφου είναι πολύ σημαντική. Οι Ευρωπαίοι ε, ποτέ κατά το παρελθόν δεν έθεσαν τόσο υψηλέ απαιτήσει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ποτέ δεν την επέκριναν τόσο δρυμή, δρυμύτατα. Ε, πρώτον, ε, όσον αφορά του πολίτε τη Ευρώπη, ε, δεν είναι δυνατόν οι πολίτε μα να αγνοούμε, δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε τις επιπτώσεις της διαρθρωτικής κρίσης όπως επίσης και όλο μεγαλύτερες προκλήσεις ε, λόγω της ε, παγκοσμιοποίησης γιατί αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά ε, αμφισβητούμε το πρόγραμμα, αυτό το project που λέγεται Ευρώπη. Αυτά λοιπόν πρέπει σαφώ να ληφθούν υπόψη στην ε, διαμόρφωση του επόμενου πολιτού σε δημοσιονομικού πλαισίου έτσι ώστε η Ευρώπη να γίνει περισσότερο κατανοητή και να στηριχθεί. Δεύτερον, η αποδοχή θα πρέπει να υπάρχει τόσο σε επίπεδο πολιτών όσο και σε επίπεδο κρατών μελών διότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός ας μην ξεχνάμε ότι παράγει υπεραξία. Και τρίτον ε, πρέπει να ε, δεχτούμε τις σκέψεις εκείνες ε, που λένε ότι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο σχετίζεται με τη στρατηγική του 2020 ως εκ τούτου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ενδεχομένω και το στοιχείο της ενότητας του προϋπολογισμού αυτού. Ο συνάδελφος Γιάνν Ολμπριχτ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι. κάποιος που δεν γνωρίζει πολλά από αυτά που συμβαίνουν μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι ανεύθυνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνοντας αύξηση του προϋπολογισμού. Θέλω όμως να ξεκαθαρίσω ότι η δουλειά της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ ήταν πολύ επικεντρωμένη, επικοδομητική και ρεαλιστική. Στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ συζητήσαμε το πόσο θα μας κοστίσουν οι πολιτικές αποφάσεις μην ξεχνάμε ότι τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών που στέλνουν κάποιες επιστολές συμφώνησαν στους στόχους της στρατηγικής του 2020. Η Επιτροπή Σούρε ε, προσπάθησε να επισημάνει το κόστος που θα έχουν οι κοινέ πολιτικές αποφάσεις. Τις αντιμετωπίζουμε με μεγάλη σοβαρότητα αν τα κράτη-μέλη αποφασίσουν να κινηθούν και εμείς οι εκπρόσωποι των πολιτών μας συμφωνούμε, τότε πρέπει να έχουμε και τα απαραίτητα μέσα για να τα πετύχουμε αυτά. Η έκθεση που θα τεθεί σύντομα σε ψηφοφορία ε, είναι μια έκθεση που έχει σωστά μελετηθεί και στηρίζεται σε συμβιβασμούς. Είναι ρεαλιστική και επιπλέον είναι μια έκθεση που αποτελεί καλή βάση για το ξεκίνημα συνομιλιών. Μπορούμε σήμερα να πούμε στην αίθουσα αυτή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις ως εκπρόσωπος της Πολωνίας θέλω να πω ότι είμαι απολύτως πεπισμένος ότι η Πολωνική Προεδρία θα είναι Προεδρία που θα ξεκινήσει πολύ ρεαλιστικές συζητήσεις ακριβώς επειδή η κυβέρνησή μας είναι φιλοευρωπαϊκή. Βεβαίως οι συζητήσεις θα είναι δύσκολες αλλά και θετικές, οικοδομητικές για το μέλλον μας. Ε, αν ξεκινήσουν πραγματεύσεις, είναι έτοιμο το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ η κυρία Γιούτα Χάουγκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από ένα χρόνο η Ολομέλεια συνέστησε την ειδική αυτή επιτροπή ε, για να ασχοληθεί με το πολιτέ σε δημοσιονομικό πλαίσιο και ανέθεσε μία εντολή στην επιτροπή αυτή. Μόνο που Ακριβώς μετά από 11 μήνες η Επιτροπή ΣΕΡΕ, ΣΟΥΡΕ με συγχωρείτε, κατέθεσε το πόρισμά της. Η δουλειά της Επιτροπής ε, χαρακτηρίστηκε από πειθαρχία και αυτό μπορούσε να γίνει μόνο αν επικρατούσε ειλικρίνεια, αλληλεγγύη και ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που συμμετείχαν στις εργασίες της Επιτροπής. Ε, έχουμε λοιπόν την έκθεση. Ε, η έκθεση αυτή κατά την άποψή μας είναι πολύ καλή γιατί πράγματι και επιμένω σε αυτό είναι μια έκθεση που αντέχει στην κριτική. Όμως για να υπάρχουν καλά αποτελέσματα δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν μόνο καλοί βουλευτές πρέπει να υπάρχουν και καλοί συνεργάτες και αυτούς τους είχαμε τους χαρήκαμε. Αυτό δεν αφορά μόνο τους ε, προσωπικούς μας ε, βοηθούς ε, και τους συνεργάτες. Οι συνεργάτες ευρύτερα περιλάμβαναν και τα μέλη της γραμματείας. Μία θαυμάσια ομάδα υπό την καθοδήγηση της κυρίας Μόνικα Στράσερα. Αυτή η ομάδα αυτή όχι μόνο ήταν επαγγελματική αλλά ενδιαφερόταν και για τη δουλειά της. Έδειξε υπομονή, δημιουργικότητα, οργανωτικότητα, ευελιξία και το καλύτερο απ' όλα, η ομάδα αυτή ήταν πάντα με καλή διάθεση. Προφανώ λοιπόν όλη αυτή η φοβερή και έντονη δουλειά του έκανε και τη χάρηκαν. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστώ εκ βάθου καρδία όλου αυτού του ανθρώπου. Uh, Von Anfang an hatten Ευθύ εξ αρχή, ο Σαλβαντόρ και εγώ είχαμε αποφασίσει να καταθέσουμε μια έκθεση η οποία θα μπορεί να στηριχθεί από τα τρία τέταρτα του Κοινοβουλίου. Μάλιστα, στην τελική ψηφοφορία επιτύχαμε ε, ε, σύμφωνη γνώμη από τα τέσσερα πέμπτα τη Επιτροπή και χαρήκαμε πολύ γι' αυτό. Εμεί ζητάμε να υπάρχει ένα πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θα στηρίζει του στόχου τη στρατηγική 2020 και παράλληλα ε, θα θέτει όλε τι πολιτικές υπό την αιγίδα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αυτό νομίζω ότι μπορείτε όλοι να το θεωρήσετε λογικό, ρεαλιστικό και εφικτό. Η δική μας η έκθεση περιλαμβάνει 174 παραγράφους, πάρα πολλά επιχειρήματα για περισσότερη Ευρώπη, γιατί πραγματικά το χρειαζόμαστε αυτό. Σας παρακαλώ, διαβάστε την έκθεσή μας. Η έκθεση αυτή αποτελεί την καλύτερη βάση για να γίνεται η συζήτηση επιτόπου με τους πολίτες και για τη συζήτηση με το Συμβουλίο, το οποίο βέβαια σήμερα λάμπει δια της απουσίας του. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή δουλειά που ε, προσφέρατε όλοι σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Άννε Και εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι η έκθεση είναι ισορροπημένη και περιέχει μια σαφή και ευέλικτη εντολή προς την Επιτροπή Προεπολογισμών που θα διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Συμφωνώ με την κυρία Ρίτα Χάγκο ότι πρέπει να τη διαβάσετε την έκθεση αυτή. Οι αρχηγοί κρατών κυβερνήσεων και υπουργοί οικονομικών βιάστηκαν να πούν ότι το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Η όλη διαδικασία ήταν πραγματικά πολύ καρποφόρα. Και συγχαίρω τον εισηγητή, συγχαίρω την ε, Κομισιόν η οποία έπαιξε πολύ δραστήριο ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Καλύψαμε όλους τους δομείς πολιτικής ε, του προπολογισμού. Η δουλειά ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι φιλόδοξο, γιατί διαθέτουμε την στατική Ευρώπη 2020 που έχει ως ε, στόχο να, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό από άλλα μέρη του κόσμου, την Κίνα και αλλού. Ε, χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ενεργειακής επάρκειας και ενεργειακής απόδοσης. Θα, μπορούσαμε, θα έπρεπε βέβαια να έχουμε και κάποιες προβλέψεις για μειώσεις ε, ε, στα διαστατικά κονδύλια, τα οποία ε, είναι επιστροφές προς τα κράτη-μέλη, ε, αλλά η έκθεση μας βοηθάει σε κάθε περίπτωση να αντιμετωπίσουμε τις καινούριες προκλήσεις και τις καινούριες προτεραιότητες, δίκτυα, ενέργεια, έρευνα κλπ. Έχουμε πλέον εν, διαπραγματευτική εντολή για να διαπραγματευτούν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και μην ξεχνάμε ότι αυτό το ποσό το οποίο προτείνουμε είναι η οροφή των δαπανών, όχι οι πραγματικές ε, δαπάνες. Ε, υποστηρίζω την έκθεση αυτή λοιπόν. Ευχαριστώ. Ε, Ο συνάδελφος Χέντεκ Φάιμον. Κυρίες και κύριοι, το, το τελευταίο διάστημα, τους τελευταίους μήνες, έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να προετοιμάσουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2020. Και θέλω να πω ένα παραμύθι του Καρλό Τσάπετ. Οι άνθρωποι αποφάσισαν να φτιάξουν μια τούρτα που να αρέσει σε όλους. Και βάλαν στην τούρτα όλα τα υλικά που υπήρχαν. Στο τέλος βέβαια τους έπιασε στο μαχόπονος φοβάμαι ότι αυτή τη μοίρα θα έχει και αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο γιατί έχουμε όλες τις υποχρεώσεις, όλες τις συστάσεις που τις έχουμε συμπεριλάβει αλλά δεν ξέρουμε αν όλα αυτά μαζί θα λειτουργήσουν. Ξέρουμε ότι απέτυχε η στρατηγική της Λισαβόνας και τώρα έχουμε τη στρατηγική του 2020. Θα θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο. Θεωρώ ότι η κλιματική αλλαγή είναι ο χειρότερος στόχος που θέσαμε. Το θέμα των ιδίων πόρων για τον προπολογισμό και ο τρόπος που θα εκδώσουμε ευρωομόλογα δεν είναι καλή λύση. Αυτό θα συνεπάγεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρεωθεί. Ο